Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Αρχίζουμε την απογευματινή μας συνεδρίαση της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης και αρχίζουμε με ψηφοφορίες. Η πρώτη ψηφοφορία που έχουμε είναι η έκθεση περιοχές που παρουσιάζουν αναπτυξιακή καθυστέρηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η κυρία Τζουφρίντα είναι η συγκεντριά μας. Μήπω θέλετε να πείτε κάτι πριν την ψηφοφορία, όχι. Καλώς. Έχουμε δύο γνωμοδοτήσεις, μία από την Επιτροπή Γεωργίας και μία από την Επιτροπή Αλίας. Όσο προχωράμε στην ψηφοφορία, θα σας πω κάποια πράγματα για την γνωμοδότηση της Επιτροπής Αλίας. Και αν δεν υπάρχει τίποτα άλλο, να αρχίσουμε να ψηφίζουμε. Συμφωνεί. Και αρχίζουμε με τροπολογία αριθμό 2. Υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχέ. Εγκρίνεται. Τροπολογία 3. Υπέρ. Κατά. Αποχέ. Εγκρίνεται. Τροπολογία 4. Υπέρ. Κατά. Αποχέ. Εγκρίνεται. 5. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 6 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 7 με προφορική τροποποίηση. Είναι κανεί κατά τη προφορική τροποποίηση, όχι. Ωραία. Ψηφίζουμε την τροπολογία 7 με την προφορική τροποποίηση υπέρ, κατά, αποχέ, εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία α. Υπέρ, κατά, αποχέ, Εγκρίνεται. Τώρα, τροπολογία 12. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 14. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβιβαστική Β. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 20. Υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 21 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 22 υπέρ, κατά, αποχές θα ελέγξουμε παρακαλώ για να δούμε τι γίνεται. Ελέγχουμε ηλεκτρονικά λοιπόν για την τροπολογία 22. Ψηφίστε. Ψηφίστε παρακαλώ. Πέρα τη ψηφοφορία. Όχι, δεν ψηφίσατε όλοι. Τι, δεν λειτουργεί. Απορρίφθηκε. Εντάξει, δεν κάνει διαφορά η μία ψήφος. Απορρίφθηκε η τροπολογία αυτή. Τροπολογία 23 τώρα. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 27 με προφορική τροποποίηση. Είναι κανείς κατά της προφορικής τροποποίησης. Όχι, ωραία. Ψηφίζουμε λοιπόν με την τροποποίηση αυτή. 27 υπέρ, κατά, αποχέ, εγκρίνεται. Συμβιβαστική γάμα. Υπέρ παρακαλώ, κατά, αποχέ. εγκρίνεται. Τροπολογία 30. Υπέρ, κατά, αποχέ. εγκρίνεται. Συμβαστική D, δέλτα, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 36 τώρα. Υπέρ παρακαλώ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 37. Α, είναι ταυτόσιμη. Είναι η ίδια με τη 36, πότε έχει εγκριθεί. 39 τώρα. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία ε τώρα. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 43. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 44. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 45. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 47. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 46 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβιβαστική F, σίγματα υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία Επιτροπής Γεωργίας, ε, άγκρι ε, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Άγκρι G, ζήτα, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Συμβαστική τροπολογία αριθμό 1. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 53. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβιβαστική 2. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβιβαστική 3. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική 3α. Υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 4 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 5 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 5α υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 6 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 7 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 7α υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 7β υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική Σ. γάμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική τρο... ε, η τροπολογία συγγνώμη 99 υπέρ κατά αποχές Νομίζω ότι εγκρίνεται. Λέει η πρόεδρος. Συμβαστική 8. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική 9. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική 10. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τώρα τροπολογία 113. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 114 υπέρ. Α, όχι. 115, γιατί 114 καταπίπτει. 115 λοιπόν τώρα υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 11 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική 11α υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 121 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 122 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 123 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 12 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 128 τώρα. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 129, καταπίπτει. Και έτσι περνάμε στη συμβαστική 13. Υπέρ, παρακαλώ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 13α. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική 13β υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβιβαστική 14 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 143 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβιβαστική τροπολογία 15 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβιβαστική 15α. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Πάμε τώρα στην τροπολογία 16 της Επιτροπής Γεωργίας. Υπέρ, κατά, αποχές, θα ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Άγκρι 16. Ελέγχουμε ηλεκτρονικά. Ψηφίστε παρακαλώ. Πέρας της ψηφοφορίας Απορρίπτεται. Τροπολογία 149 τώρα. Με προφορική τροποποίηση. Είναι κανείς κατά της τροποποίησης, όχι. Ωραία, 149. Με την τροποποίηση υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 154. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβιβαστική τροπολογία 16. Υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 17 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 18 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 18α υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τώρα βλέπετε στον κατάλογο ψηφοφορίας ότι έχουμε τώρα τις τροπολογίες της Επιτροπής Αλίας. Θα επισυνάψουμε την γνωμοδότηση της Επιτροπής Αλίας στην έκθεσή μας, οπότε τώρα περνάμε στην τελική ψηφοφορία. Τελική ψηφοφορία λοιπόν ηλεκτρονικά. Ψηφίστε παρακαλώ. πέρα στις και συγχαρητήρια στην εισηγήτρια. Εγκρίθηκε η έκθεση. Και περνάμε τώρα στην επόμενη ψηφοφορία μας που είναι η έκθεση της κυρίας Βαλίνα. Ρόλος των περιφερειών και των πόλεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην εφαρμογή της Συμφωνίας των Παρισίων COP20. Να πείτε κάτι πριν. Όχι, δεν χρειάζεται. Α, καλώς τότε. Οπότε περνάμε κατευθείαν στην ψηφοφορία. Και αρχίζουμε με την τροπολογία αριθμού 1. Υπέρ παρακαλώ, κατά, αποχές, έγκρινεται. Τροπολογία 2. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 3. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 4. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 5 υπέρ, κατά, αποχές, θα ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Για να δούμε. Η ηλεκτρονική ψηφοφορία για την τροπολογία 5. Ψηφίστε παρακαλώ. Πέρας της ψηφοφορίας και εγκρίθηκε. Πάμε τώρα στην τροπολογία 6. Δεύτερο τμήμα όμως. Γιατί κρίναμε την 5. Οπότε ψηφίζουμε το δεύτερο τμήμα της τροπολογίας 6. Υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές. Εγκρίθηκε. Τροπολογία 7 τώρα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική αριθμός 1. Υπέρ παρακαλώ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική 2. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική 3. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική 4. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 23 τώρα. Υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές. Έγκριθηκε. Συμβαστική 5. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Έγκρινεται. Τροπολογία 24. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Έγκρινεται. Συμβαστική 6. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 7 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 33 τώρα. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 35. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 35 υπέρ, κατά, αποχές, θα ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Τροπολογία 35. Μπορείτε να ψηφίσετε ηλεκτρονικά. πέρασε της ψηφοφορίας εγκρίθηκε. Α, όχι, συγγνώμη, απορρίφθηκε διορθώνει ο πρόεδρος. Απορρίφθηκε. Τροπολογία 36. Ψηφίζουμε 36 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Θέλετε να ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Ωραία. Ελέγχουμε για την τροπολογία 36 ηλεκτρονικά. Ψηφίστε παρακαλώ. Πέρα της φοφορίας εγκρίθηκε. Τροπολογία 37 τώρα. Μάλλον 38. 38 διορθώνει ο πρόεδρος. 38. Υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές. Για να ξαναψηφίσουμε παρακαλώ υπέρ. Κατά. Αποχές. Έγκρινεται νομίζω. Να ελέγξουμε. Καλώς. 38. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. Μπορείτε να ψηφίσετε. Πέρα της ψηφοφορίας. Εγκρίθηκε. Τώρα, συμβιβαστική 8. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 45. Σωστά. Ναι, 45. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 46. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Συμβαστική 9. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική 10. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 54. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 55. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 56. Υπέρ, καταπίπτει εντάξει, και η 57. Οπότε πάμε στη συμβαστική. Συγγνώμη, λέει πρόεδρος. Η 57 είναι μια τροπολογία που πρέπει να ψηφίσουμε. Ποιοι είναι υπέρ της 57 λοιπόν, παρακαλώ. Κατά, αποχές εγκρίνεται. Τώρα πάμε στη συμβαστική 11. Υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 12 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβιβαστική 13 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 65 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 66 υπέρ, κατά, διακοπή εκτός μικροφώνου. Ήμασταν στην 65 και 66. Αυτό έχω εγώ μπροστά μου και δεν φαίνεται ότι καλύπτονται από τις συμβαστικές. Φαίνεται κυρία Κρέλα ότι έχετε δίκιο, ότι ο δικός μου κατάλογος δεν είναι σωστός. Αυτό τι σημαίνει, ότι πρέπει να ψηφίσουμε ενώ είναι στη συμβαστική. Εντάξει, το διασκεδάζουμε σήμερα στη ψηφοφορία. Τι να κάνουμε. Λυπάμαι. Πάμε πίσω, λοιπόν. Τροπολογία 65. Υπέρ, παρακαλώ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 66. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 67. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται νομίζω, αλλά σε ελέγξουμε καλύτερα ηλεκτρονικά για την 67. Μπορείτε να ψηφίσετε. Τέλος, απορρίφθηκε. Τροπολογία 68. Καταπίπτει. Αν εγκρίναμε την 67, αλλά δεν την εγκρίναμε. Οπότε 68. Ποιοι είναι υπέρ? κατά, αποχές, εγκρίνεται. 69 αυτή καταπίπτει. Γιατί εγκρίναμε την 68. Ωραία. 70 όχι. Δεν καταπίπτει. Ωραία. 70 υπέρ παρακαλώ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 14. Θέλετε να ελέγξουμε για την 70 ηλεκτρονικά. Ωραία. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. Ψηφίστε παρακαλώ. Τέλος. Απορρίπτεται. Τώρα συμβαστική 14. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 74. Τώρα. Υπέρ παρακαλώ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 75. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 76. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Να ελέγξουμε ηλεκτρονικά για την 76 καλύτερα. Ψηφίστε παρακαλώ. Τέλος. Εγκρίθηκε. Συμβαστική 15. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβιβαστική 16. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 89 τώρα. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 90. Υπέρ, κατά, αποχές, το ίδιο, απορρίπτεται. Θέλετε να ελέγξουμε για την 90. Ωραία. Η ηλεκτρονικά ψηφίζουμε λοιπόν για την 90. Ψηφίστε. Τέλος. Εγκρίθηκε. Εγώ έφταιγα. Λάθος μου. 91 καταπίπτει εφόσον εγκρίθηκε 90. 92 τώρα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 93. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίθηκε. 99. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική 17 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 108 τώρα. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική 18 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική 19 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβιβαστική 20 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική 21 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβιβαστική 22 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβιβαστική 23 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική 24 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβιβαστική 25 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 116 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Τροπολογία 117 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 118 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται νομίζω. Να ελέγξουμε. Κατά, αποχές, εγκρίνεται. Και τώρα περνάμε στην ψηφοφορία της τροποποιημένης έκθεσης ηλεκτρονικά. Μπορείτε να ψηφίσετε. τροποποιημένης έκθεσης ηλεκτρονικά. Μπορείτε να ψηφίσετε. Πέρας της ψηφοφορίας και εγκρίθηκε η έκθεση. Συγχαρητήρια στην εισηγητρία. Και να τη θυμόσαστε αυτή τη ψηφοφορία με τα λάθη που έκανα, λέει η πρόεδρος. Και τώρα συνεχίζουμε και περνάμε στην γνωμοδότησή ε, μας για το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο για τον συντονισμό των οικονομικών πολιτικών. της Επισκόπης Ανάπτυξης για το 2018. Εγώ είμαι η συγκήτρια. Και ξεκινάμε με την ψηφοφορία. Λοιπόν, συμβαστική 1 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται.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 Εγκρίνεται και τώρα μπορούμε να ψηφίσουμε για το σύνολο. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας, εγκρίνεται η έκθεση. Σας ευχαριστώ. Και η τελευταία για σήμερα για την υλοποίηση του Γενικού Προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το, έτος, για το οικονομικό έτος 16 Εγώ είμαι η συγγήτρια, θα πάμε απευθεία στην ψήφο. Συμβαστική λοιπόν ένα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 13 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 4 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Σημαστική 5 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 20 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 21 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 6 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 25 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 7 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 32 υπέρ 32 λέμε υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 33 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 34 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 8 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Και πάμε στην τελική ψήφο Άρχεται η ψηφοφορία, παρακαλώ. πέρα τη ψηφοφορία και εγκρίνεται η έκθεση. Σας ευχαριστώ πολύ. Και σας ευχαριστώ και για την υπομονή σας με, την, ε, με τις σημερινές ψηφοφορίες, τις οποίες ολοκληρώσαμε και μπορούμε να προχωρήσουμε στο επόμενο σημείο της μεσίας Διατάξεως. έχουμε ανταλλαγή απόψεων Thank Με την κυρία Ιβάνοβα, που είναι μέλος του Ελεκτικού Συνεδρίου, σχετικά με το έργο του συνεδρίου στον τομέα της πολιτικής συνοχής. Η κυρία Ιβάνοβα έχει ξαναέρθει στην Επιτροπή μας, είχαμε τη χαρά σήμερα ως συνήθως θα δώσω το λόγο στην κυρία Ιβάνοβα για μια αρχική τοποθέτηση και μετά στα μέλη ξεκινώντας από τους συντονιστές. Έχουμε χρόνο, θυμίζω, μέχρι αξιότιμα μέλη. Πάντα με χαρά έρχομαι εδώ στην Επιτροπή Ρέτζι και ευχαριστώ για την πρόσκληση. Το συζητούσαμε από πέρυσι αυτό το ελεγκτικό συνέδριο αφιερώνει σημαντικό τμήμα της δουλειάς του στην πολιτική συνοχή, όχι μόνο στα πλαίσια της ε, ετήσιας έκθεσης, αλλά και διαφόρων εκθέσεων επίδοσης. Και αυτά που είχα σκεφτεί σήμερα να συμπεριλάβω, μάλλον υπάρχουν τόσο, τόσα πολλά σημαντικά ως προς την πολιτική συνοχή δηλαδή. ξεκινώ από την συμμόρφωση και δεν ξέρω αν λειτουργεί το σύστημα με τις διαφάνειες. Εδώ σε αυτό το γράφημα που είναι αρκετά απλό μπορείτε να δείτε που δείχνει μια αύξηση του ρυθμού αλλά και 10 χρόνια νωρίτερα να πάμε τα ποσοστά λάθους ήταν διψήφια. Είχαμε και 11 ακόμα τις 100 στην προηγούμενη προγραμματική περίοδο, το 5,7% στο 4,8% μέχρι το 2016. Βεβαίως πρέπει ακόμα να σημειώσω ότι όλα αυτά βεβαίως είναι πάνω από το όριο, το κατόφλι που είχε οριστεί στο 2%. Επομένως είναι μία από τις περιοχές πολιτικής που μαζί με την πολιτική γεωργίας είναι υψηλή. Το σφάλμα δεν σημαίνει παραβίαση ή απάτη ή κατασπατάληση. Μιλούμε για σφάλματα διαφόρων ειδών συμπεριλαμβανομένων διοικητικών σφαλμάτων, λανθασμένες ημερομηνίε στις, ε, στα έντυπα που υπευλήθησαν Πάνια. Θα προσπαθήσω να σας ε, παρουσιάσω τους πιο συνηθισμένους τύπους ήδη λαθών, σφαλμάτων, στις προμήθειες έχουμε πάρα πολύ συχνά μια σημαντική πηγή. Μαζί με τις δηλώσεις δαπανών 42% συνολικά των σφαλμάτων. Πάντα οι προμήθειες είναι στο top 3. Και εδώ βλέπουμε στο 30% μαζί με μία επιλέξιμη δραστηριότητα ελέγχοντας τις συναλλαγές 135 από τις 1.437 έχουν χρησιμοποιήσει απλουστευμένες επιλογές υπολογισμού, κόστους δηλαδή, και εκεί όπου βλέπουμε την απλούταση ε, να γίνονται σφάλματα. Στην επόμενη διαφάνεια ήθελα σύντομα απλώς να αναφερθώ σε κάποιες πτυχές ενός στοιχείου που έχουμε την πρόθεση να αλλάξουμε για του χρόνου σχετικά με ποιο τρόπο, με ποια μεθοδολογία υπολογίζαμε, αξιολογούσαμε την αξιοπιστία των δεδομένων. Βεβαίως έχουν γίνει τροποποιήσεις στο νομοθετικό πλαίσιο όπως η ετήσια διαδικασία ελέγχου μαζί με το 10% της παρακολουθίας για τις δηλώσεις του 2017 θα προσπαθήσουμε να μετακινηθούμε από την παραδοσιακή προσέγγιση για τον έλεγχο νομιμότητας προς την καλύτερη χρησιμοποίηση έργου που και αν είναι θα μπορέσουμε να πάμε προς αυτό που ονομάζουμε δήλωση εγγύησης το οποίο θα μας επιτρέψει μια σειρά από ωφέλη για αρκετά χρόνια μας διευκολύνει τα κρατη γιατί θα μπορέσουμε να παρέχουμε μεγαλύτερο επίπεδο λεπτομερίας. Βεβαίως η μείωση του διοικητικού άκθους για τους δικαιούχους είναι πολύ σημαντική. Πολύ συχνά ακούμε ότι ένας δικαιούχος μπορεί να ελεγχθεί όχι μία και δύο άλλα διοικητικό άκθος. Με την προσέγγιση λοιπόν αυτή θα βοηθήσουμε και τους δικαιούχους. Αυτά είναι συντομία για τα στοιχεία συμμόρφωσης, που είναι μόνο μία πτυχή της νομότητας. Δεν είναι το σύνολο. Και έχει ενταχθεί, αν θέλετε, στο νέο πνεύμα του επομένου πουδουπού πολιετούς δημοσιονομικού πλαισίου, για διάφορες πτυχές αποτελεσματικότητας επίδοσης και αποτελεσμάτων δηλαδή της υλοποίησης της πολιτικής νοχής. Και εδώ προσπαθώ να απεικονίσω είχε πλήρως μερικός ή όχι τους στόχους τους. Ε, ε, βλέποντας κανείς τα μεγέθη το 58% βλέπουμε ότι έχει πετύχει. Γραμμίζονται με τα επιχειρησιακά προγράμματα των έργων δηλαδή ώστε να έχουν επιτύχει τους στόχους τους και ε, σε όλα τα χρόνια βλέπουμε με συγκεκριμένη εστίαση ή θέμα για την πολιτική μεταφορών, για το δικό δίκτυο, για τα εσωτερικά ε, πλωτά και από άλλους συναδέλφους του τμήματος 2 για τους άξονες προτεραιότητας ε, μετα... όχι υψηλής προτεραιότητας αλλά πάντοτε προτεραιότητας που όχι όλες από τις στοιχείες αυτές δεν είναι σχετικές δηλαδή για την ε, Επιτροπή σας αλλά η διάρκεια των έργων, η ταχύτητα των δικτύων, η απορρόφηση, η βιωσιμότητα και κάτι που δεν είναι ακριβώς δεν εμπίπτει ακριβώς το θέμα, αλλά ε, σκέφτηκα ότι θα ήταν καλό να το αναφέρω σχετικά με την γνωμοδότηση του συνεδρίου για τις προτάσεις του επομένου ε, πολιετούς δημοσιονομικού να υπογραμμίσει κανείς τα βασικά μηνύματα του ενημερωτικού αυτού εγγράφου. Καταρχάς, και το πιο σημαντικό, είναι να καθορίζεται σωστά η προσθεθέμενη αξία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Να αναπτυχθεί δηλαδή ένα σκεπτικό που και μεγαλύτερη ή πιο συγκεκριμένη απόδοση ευθυνών σε περίπτωση που υπάρχουν να δείτε σε μεγαλύτερη λεπτομέρεια σε τι συνίσταται αυτή η νέα προσέγγιση. Αυτή ήταν η πρώτη μου τοποθέτηση. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ θα χρησιμοποιήσουμε αυτή την ευκαιρία που μας δώσατε να προσκαλέσουμε συναδέλφους σας για κάποια από τις εξειδικευμένες εκθέσεις που έχει συντάξει το ελεγκτικό συνέδριο και φυσικά σας ευχαριστούμε πολύ που μας υπενθυμίσατε Ναι, γιατί είμαι πάρα πολύ χαρούμενος. Είναι να γίνουμε πιο αποτελεσματικοί, να, να δουλεύουμε καλύτερα να βελτιώσουμε την νομοθεσία μας ώστε τα κράτη-μέλη, οι περιφέρειες, οι δήμοι να έχουν χαμηλότερα ποσοστά ασφάλματος. Και φαίνεται αυτή η φθήνουσα πορεία του ποσοστού σφάλματος που ε, το να υπήρχαν πολλά σφάλματα θα έστελνε λάθος μήνυμα. Και όπως είπατε είναι σημαντικό να αποδίδεται εμπιστοσύνη και να υπάρχει εμπιστοσύνη εκεί που χρειάζεται. Και είναι σημαντικός παράγοντας η εμπιστοσύνη για την επόμενη προγραμματική περίοδο και το βασικό μας ε, ε, αίτημα είναι να απλουστευτεί η διαδικασία, να μην υπάρχουν τόσα πολλά ασφάλματα. Λοιπόν, εγώ ε, έχω λάβει την, την έκθεση αυτή, βλέπω ότι Το Jasper λοιπόν είναι ένα από τα τρία προγράμματα J. Και σκοπός αυτού του προγράμματος του Jaspers είναι να βοηθηθούν τα κράτη-μέλη. Βεβαίως ε, ε, επικεφαλής ε, είναι η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων που υποστηρίζει αυτά τα μεγάλα έργα από την προηγούμενη προγραμματική περίοδο. Όταν λοιπόν, καθώς παρακολουθούσα την παρουσίαση, είχα πάρα πολλές ανησυχίες και αμφιβολίες για το πώς ακριβώς γίνεται η διαχείριση, η διεύθυνση αυτού του, του, του προγράμματος. Αφενός δηλαδή τα, τα, τα, κράτη-μέλη είναι αυτά που ε, δίνουν τα χρήματα, ταυτόχρονα είναι και εκείνα που παραλαμβάνουν το, τα χρήματα. Το, όλα μέσα σε ένα, σε, σε, σε ένα πλαίσιο, μέσα σε ένα γραφείο και μόνο, ε, το οποίο όλο και αυξανόταν ως προς το προσωπικό του, Φαινόταν λοιπόν να υπάρχει μια αντιφατική πορεία από άποψη όγκου αφενός εργασίας και αφετέρου του, του όγκου των έργων που χρηματοδοτούνταν. Νομίζω ότι πρέπει να, να πάρουμε μια απόφαση. Αν θέλουμε να συνεχίσουμε αυτό το project, το Jaspers, με τεχνική συνδρομή και ιδίως για τα νέα κράτη-μέλη. Αν όμως φαίνεται ότι δεν αποφέρει τα επιθυμητά αποτελέσματα Γι' αυτό παραμένει ανοιχτό με ερωτηματικό εμπάση περιπτώσει στην έκθεση. Αν δηλαδή τελικά καταλήγει αυτό το project να, να βοηθάει όλα τα έργα χωρίς να υπάρχει κάποια ιεράρχηση, ε, δεν ξέρω αν έχει νόημα να συνεχίσουμε. Εξαίρετε εσείς κάτι παραπάνω ή δεν έχετε ενημέρωση. Λοιπόν, θέλω να πω και ιδιαίτερο αυτή η προφορία. Πιο πολύ ακόμα με ικανοποιεί το γεγονός ότι εκεί που χρησιμοποιήθηκε η ε, απλουστευμένη επιλογή κόστου έγιναν ακόμα λιγότερα ασφάλματα. Γιατί αυτό δίνει τον, το μήνυμα, στέλνει το σήμα ότι ε, η απλούστευση ε, στην πολιτική συνοχή είναι ο σωστός δρόμος για να προχωρήσουμε. Τα τελευταία χρόνια ε, έχω την αίσθηση ότι τα σφάλματα στην πολιτική συνοχής οφείλονται στο πολύ περίπλοκο σύστημα κανόνων και γραφειοκρατίας που έχουμε θεσπίσει. Ελπίζω λοιπόν ότι θα υπάρχει ε, υψηλή ποιότητα στην πολιτική συνοχή στο μέλλον, αλλά με απλουστευμένες διαδικασίες, κάτι που θα οδηγήσει σε σημαντική μείωση των σφαλμάτων στην πολιτική συνοχή. Και αυτό είναι ένα ε, θετικό μήνυμα ε, όχι μόνο για εκείνου που ασχολούνται με όλες αυτέ τις γραφειοκρατικέ διαδικασίες αλλά και εκείνου που δυστυχώς ε, επηρεάζονται από τον κίτρινο τύπο όπως είναι η εφημερίδα Bild στη Γερμανία η οποία διαρκώς βγάζει θέματα ότι λόγω της πολιτικής συνοχής κατασπαταλώνται εκατοντάδε εκατομμύρια στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αυτό είναι πολύ θετικό. Έχω ένα ερώτημα, μπορεί να παρεξήγησα, αλλά είπατε κάποια στιγμή ότι υπήρχαν σφάλματα κάτι σε σχέση με, με, με συμφωνίες εταιρικής σχέσης. Μπορείτε να μου το ξαναεξηγήσετε γιατί δεν κατάλαβα ακριβώς. Μιλήσατε για συμπράξεις δημοσίου-ιδιωτικού τομέα. Ίσως, ίσως παρεξήγησα, ίσως να παρανόησα. Δεν, δεν κατάλαβα τι σχέση έχει αυτό που είπατε με το ελεγκτικό συνέδριο. Σας ευχαριστώ. Ωραία, ευχαριστούμε πολύ. Η κυρία Τόμασίτς Θέλετε το λόγο, όχι. Εντάξει. Δεν βλέπω τους άλλους συντονιστές. Ξεκινάμε λοιπόν με τα μέλη της Ρέτζη. Ο κύριος Μπούντα έχει το λόγο. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ κυρία Ιβανόβα για την παρουσίασή σας. ότι είναι, ο μεγαλύτερος εχθρός θεωρούν ότι είναι το ελεγκτικό συνέδριο. Δυστυχώς. Ε, εγώ, ξέρετε, κατάγομαι από τη Ρουμανία και μου λένε οι ψηφοφόροι. Φοβούνται οι άνθρωποι ότι μετά πρέπει να, ενδέχεται να, να, να πρέπει να ξεπληρώσουν, ε, να ξαναπληρώσουν, να, να επιστρέψουν χρήματα πέσουν τα χρήματα αυτά, φυσικά πού να τα βρουν αυτά τα χρήματα, τα έχουν ήδη επενδύσει, έχουν ήδη φύγει αυτά τα χρήματα. Θέλω να πω ότι είναι πραγματικά σημαντικό τα ευρωπαϊκά ταμεία να διέπονται ανώνες των ταμείων και τι θα πει το ελεγκτικό συνέδριο και όλα αυτά. Με, με άλλα λόγια, θέλω να πω καλύτερα να υπάρχει μια καλύτερη διαβούλευση, μια ενεργή συμμετοχή. Ότι υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα. Γιατί αν εδώ στι Βρυξέλλε υπάρχουν δύο και τρει προποθέσει στο πλαίσιο τη αρεσιμότητα που μπορεί να δημιουργούν εμπόδια, φανταστείτε τι γίνεται στη... την παρουσίασή σα. Βλέπουμε για άλλη μια φορά ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των σφαλμάτων εμφανίζονται στις δημόσιες προμήθειες και φυσικά τη, τη μη επιλεξιμότητα έργων και δικαιούχων, αλλά στις δημόσιες προμήθειες. Θα ήθελα να μου πείτε αν έχετε περισσότερο ε, μιλούμε για τον, ε, για τον δημόσιο τομέα, για δημόσιες φορείς. Γιατί ε, αμφότεροι ε, δεσμεύονται από τους κανόνες για τις δημόσιες προμήθειες. Αν μιλούμε για ιδιωτικούς φορείς όμως, ίσως θα πρέπει να, να αυτό που είπατε για την πτυχή της επίδοσης, της αποτελεσματικότητας, ότι υπάρχει έλλειψη κατάλληλων κριτηρίων ε, που να θεσπίζονται στην αρχή ε, της εκτέλεσης ενός έργου. Αυτό σημαίνει ότι οι δείκτες που έχουμε είναι μη ρεαλιστικοί, και ότι δεν χρησιμοποιούνται καν δίκτες κατά την εναρκτήρια φάση υλοποίησης ενός έργου. Επίσης για τις παραβάσεις κόστους. Αυτό είναι κάτι που θα μπορούσε να είναι πάρα πολύ επικίνδυνο στο βαθμό που λέω τίμημα και συνέχεια να γίνεται μια παράβαση του κόστους, μια υπερκοστολόγηση. Ε, θέλω να μου εξηγήσετε τι ακριβώς συμβαίνει στην πράξη με αυτή την περίπτωση. Ευχαριστούμε πολύ για τις ερωτήσεις αυτές. Η κυρία Ιβάνοβα τώρα θα απαντήσει στο όλους για τις πολύ ενδιαφέρουσε ερωτήσεις σας. Θα προσπαθήσω να απαντήσω με τη σειρά που τις θέσατε. Στον κύριο Φανίστερο η πρώτα. Σας ευχαριστώ για την ερώτησή σας και σας ευχαριστώ και για τα θετικά σας λόγια όσον αφορά το στόχο, να δουλέψουμε καλύτερα και να ε, προσφέρουμε αποτελέσματα όσον αφορά την πολιτική συνοχής. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας για το ότι οι επιδόσεις βοηθούν να υπάρξει εμπιστοσύνη. Η απλούστευση επίσης. Όσον αφορά την έκθεση για το Γιάσπερ, ο Όσκαρ Χέριξ, ο συναδερφό μου, είναι υπεύθυνο και νομίζω ότι έχετε ήδη επαφή μαζί του. Του έχετε ζητήσει περισσότερε λεπτομέρειε, Πράγματι, είναι ιδιαίτερα επικριτική η έκθεση. Συστήνουμε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή διάφορε δράσει που θα έπρεπε να αναλάβει προκειμένου να ελέγξει περισσότερο το στον στρατηγικό σχεδιασμό πρώτα απ' όλα του Γιάσπερ ε, και πώς ε, σταδιακά θα εξαφανιστεί άπαξ και ο στόχο έχει επιτευχθεί Μιλάμε για έλλειψη αμεροληψίας. Γι' αυτό και προσφέρουμε ε, συμβουλευτική και βοήθεια βάσει των προγραμμάτων ε, που περιλαμβάνονται μέσα στο Γιάσπερς. Πρέπει επίσης η δυνατότητα οικοδόμησης ικανοτήτων να προσαρμοστεί, ώστε ανεπώς που είναι ο υπεύθυνο για την έκθεση αυτή θα μπορέσει να σας δώσει περισσότερες λεπτομέρειες όταν θα έχετε επαφές μαζί του. Για την κυρία Κρέλ τώρα. Πράγματι, όπως είπατε, το επίπεδο σφάλματος έχει μειωθεί και οι δυνατότητες που έχουν και που χρησιμοποιούν πιο απλοποιημένες μεθόδους. Βλέπουμε ότι σχεδόν δεν υπάρχουν πια σφάλματα. Αυτό δείχνει λοιπόν ότι όταν χρησιμοποιούνται τα αποτελεσματικά μέσα που διαθέτουμε είναι πολύ καλύτερα. Την περιπλοκότητα. Εδώ και 10 χρόνια γίνεται αυτή η συζήτηση. Υπάρχει η ομάδα υψηλού επίπεδου και το έγγραφο που ετοιμάζουμε στο ελεγκτικό συνέδριο είναι ακριβώς έχει ακριβώς ως στόχο να αξιολογήσουμε ό,τι έχει γίνει μέχρι τώρα και να παρουσιάσουμε μια επισκόπηση όλων των προτάσεων προκειμένου να σας βοηθήσουμε εσάς να παίρνετε καλύτερες αποφάσεις. Εδώ όμως θα ήθελα να αναφέρω και τη σημασία που έχει η μέτρηση των καλοπραγμάτων γιατί δεν ξέρω για την εταιρική σχέση υπάρχει βέβαια σχέση δημοσίου ιδιωτικού τομέα έτσι αλλά υπάρχει και η εταιρική συμφωνία που είναι κάτι διαφορετικό. Αυτή είναι μια έκθεση που έχει ήδη δημοσιεύσει το ελεγκτικό συνέδριο και είναι και πολύ σημαντική. Γιατί αναφέρεται ακριβώς στο θέμα της απλούστευσης, ότι μερικές φορές έχουμε υπερβολικά πολλούς δείκτες που βαραίνουν υπερβολικά τη διαδικασία, όχι μόνο το τελικό δικαιούχο, αλλά όλους όσοι συμμετέχουν στη διαδικασία δημιουργούνται χιλιάδες δείκτες σε περιφερειακό επίπεδο, σε κάθε επίπεδο που μπορεί να σκεφτεί κανείς για να μετρήσουμε τα πάντα. Μερικές φορές ακόμα και πράγματα που δεν χρειάζεται να τα μετρήσουμε. Και τελευταία είναι πολύ δύσκολο στο τέλος να έχουμε μια το έχουμε ένα συμπέρασμα που να έχει νόημα. Αυτό λοιπόν που συστήνουμε στην έκθεσή μας είναι να σταματήσει η χρήση των ε, άχρηστων δικτών. Μετρούν μεν κάτι, αλλά τελικά δεν μας βοηθούν να μετρήσουμε μια επίδοση, το αποτέλεσμα. Και ακριβώς εδώ είναι που πρέπει να κάνουμε τη διαφορά ανάμεσα στην μέτρηση αυτού που έχουμε τελικά και στην μέτρηση του πραγματικού αποτελέσματος της επίδοσης. αν μετρήσετε. Πίπτωση που έχει αυτό, δηλαδή αφού φτιαχτεί ο δρόμος, να δούμε. Έχει μειωθεί η κυκλοφοριακή συμφόρηση, είναι πιο μάνετη η κυκλοφορία, εξυπηρετείται περισσότερος κόσμος. Αυτό μας ενδιαφέρει, όχι απλώς το ξεκάθαρο αποτέλεσμα. Βλέπουμε κάποια περιφερειακά αεροδρόμια, τα οποία δημιουργήθηκαν, αλλά δεν χρησιμοποιούνται για το σκοπό που δημιουργήθηκαν. Αυτό πρέπει να έχουμε υπόψη μας λοιπόν. Είναι ξεκάθαρο. Κύριε Μπούντα, ε, λυπάμαι που σας άκουσαν πολύ έλεγχοι. Βαραίνουν την διαδικασία, την κάνουν πιο δύσκολη. Το αναγνωρίζω και το είπα και στην αρχή ότι αυτό είναι ένας από τους λόγους για τους οποίους θέλουμε να αλλάξουμε την προσέγγισή μας όσον αφορά την αξιολόγηση των παρατυπιών και αυτό πιστευτούμε τη δουλειά που κάνουν οι άλλοι βέβαια, τότε το επίπεδο ελέγχων θα είναι χαμηλότερο. Από την άλλη, δεν μπορούμε να καταλήψουμε και τους ελέγχους, γιατί είμαστε υπεύθυνοι, λογοδοτούμε απέναντι στον Ευρωπαίο Φορολογούμενο για την κάθε δεκάρα. Οπότε αυτό... Ε, κυρία Λέτης, εσείς αναφερθήκατε στα σφάλματα των ε, δημοσίων προσφορών. Εδώ ε, δεν κάνουμε διάκριση. Τυχαία διαλέγουμε, μπορούσε να είναι στον ιδιωτικό τομέα, στο δημόσιο. Όχι πολύ πρόσφατα, αλλά έχουμε μια ειδική έκθεση για τις δημόσιες προσφορές, τις δημόσιες προμήθειες. Αν θέλετε περισσότερες πληροφορίες, πιο συγκεκριμένα στοιχειούχους ιδιωτικού δημόσιου τομέα. Και για τους δείκτες, νομίζω ότι ήδη απάντησα. Αυτά. Πρόεδρο, σε ευχαριστώ. Ο κύριος Μπούντα θέλει κάτι να προσθέσει. Ναι, ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Θέλω όντω να κάνω μια διευκρίνηση. Εγώ δεν είπα ότι το ελεγκτικό συνέδριο είναι ο εχθρός μας και ότι εμποδίζει την απορρόφηση των κονδυλίων. Ούτε οι ούτε τίποτα. Το ελεγκτικό συνέδριο αντίθετα προσπαθεί να διευκρινίσει, να μου απαντήσετε στο εξή. Γιατί συχνά με ρωτάνε στη χώρα μου. Γιατί υπάρχει μια τόσο διαφοροποιημένη διαδικασία απορρόφησης των ευρωπαϊκών κονδυλίων είναι διαφορετικά τα πράγματα από τη μία χώρα στην άλλη. Γιατί στην Πολωνία, α πούμε, με ρωτάνε, ή σε αυτό δεν μου απαντήσατε. Εγώ πιστεύω ότι σε αυτό πρέπει να παρεύουν οι Βρυξέλλες. Πρέπει να υπάρξει ένα μηχανισμό που να απλοποιεί την απορρόφηση από πλευρά των χωρών μελών. Ο κόσμο κυκλοφορεί στην Ευρώπη και μαθαίνει τι συμβαίνει στη μία χώρα και στην άλλη. Εξού και δυσαρέσκεια στη συνέχεια. Και όσον αφορά το ελεγκτικό του κανόνε από ό,τι άλλε χώρε. Και γι' αυτό και δικαιούχοι στη συνέχεια έχουν δυσπιστία και επιφυλάξει. Ευχαριστούμε, ναι. Εντάξει, η κυρία Βάναβα να απαντήσει. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας αυτό που λέτε. Γιατί είναι τόσο δύσκολη η απορρόφηση, δεν ξέρω. Αν δεν την ακούσατε μέχρι τώρα, δεν είμαι σε θέση σε ένα λεπτό να σας τη δώσω. Όμως, ίσως, βρείτε μερικώς τουλάχιστον απαντήσεις στην επερχόμενη εκθεσή μας για την απορρόφηση. Γιατί τους επόμενους μήνες θα Πάντως, άπαξ και δημοσιευθεί η έκθεση αυτή, φαντάζομαι να βρείτε εκεί κάποιες από τις απαντήσεις που ψάχνετε. Πρόεδρος, ωραία κύριε Ιβάνοβα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Δεν έχουμε άλλες ερωτήσεις. Κάτι το οποίο για μένα δείχνει ότι όσε πολλές ερωτήσεις να σας κάνουμε. Τώρα, επειδή βρισκόμαστε τακτικά, η επικοινωνία μας βοηθάει και υπάρχει περισσότερη εμπιστοσύνη. Σας ευχαριστούμε πολύ και ευχαριστούμε που απαντήσατε στις ερωτήσεις μας. Θα συνεχίσουμε τις επαφές και τη συνεργασία με το ελεκτικό συνέδριο. Ωραία, τώρα αγαπητοί, πέντε. Οπότε σας παρακαλώ, πέντε ακριβώς να είσαστε εδώ.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 Πάλι Ευχαριστώ.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 Good afternoon, ladies and gentlemen, again. After the short break, I have a... Μετά από αυτή τη ε, διακοπή, καλωσορίζουμε τον προσκεκλημένο μας, τον κύριο Ντομπρόσκης, Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αρμόδιο για το ευρώ και τον κοινωνικό διάλογο, επίσης υπεύθυνο για τη χρηματοπιστική σταθερότητα, τις χρηματοπιστικές υπηρεσίες και την Ένωση Κεφαλαίου Αγορών. Η ανταλλαγή απόψεών μας θα επικεντρωθεί στο πρόγραμμα στήριξης διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και την υλοποίηση αυτού. Όπως θα θυμάστε, η Επιτροπή Ρέτζι ήταν αρμόδια για το νομοθετικό φάκελο, για την ε, θέσπιση, τη δημιουργία αυτού του προγράμματος και σε τακτά χρονικά διαστήματα ενημερωνόμαστε από την Επιτροπή σχετικά με τις εξελίξεις γύρω από αυτό το πρόγραμμα. Σας ευχαριστούμε πολύ. Και στο τέλος του 2017 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε μια νομοθετική πρόταση για την, για τον, για την ενισχυμένη Οικονομική και Νομισματική Ένωση. Μία από αυτές τις ε, ε, νομοθετικές προτάσεις για, την, για τις οποίες η Επιτροπή μας είναι ε, υπεύθυνη είναι η ενίσχυση του SRSP και τη δημιουργία ενός νέου προγράμματος για την ενίσχυση της σύγκλησης στην Ευρωζώνη. Σήμερα λοιπόν έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε όλα αυτά τα θέματα με τον κύριο Ντομπρόσκης και για να μην χρονοτριβήσουμε περαιτέρω θα του δώσω το λόγο και στη συνέχεια θα γίνει συζήτηση με τα μέλη της ε, Επιτροπής. Αξιότιμα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, καταρχάς να σας ευχαριστήσω για την πρόσκληση που μου απευθύνατε και τη δυνατότητα να συζητήσουμε αυτό το πρόγραμμα στήριξη διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων όσον αφορά τον σχεδιασμό, την υλοποίηση και την αξιολόγηση ε, των μεταρρυθμίσεων και την, ε, με σκοπό την καλύτερη και αποτελεσματικότερη χρήση των ε, ενωσιακών και συγκεκριμένα των διαρθρωτικών ταμείων. Οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις είναι πολύ σημαντικές για την συνοχή, τη σύγκληση και την χωρίς διακρίσεις ανάπτυξη. Είναι απαραίτητο στοιχείο μιας σύγχρονης οικονομία βοηθά στις επενδύσει και τη δημιουργία θέσεων απασχόληση. Επίση, οι μεταρρυθμίσει μειώνουν τις ε, διαρθρωτικές ε, ανισορροπίες και ανισότητες μεταξύ ευρωπαϊκών χωρών και περιφερειών. Το SRSP συμβάλλει ε, ενισχύοντας διοικητικές ανισορροπίες και ανισότητες μεταξύ ευρωπαϊκών χωρών και περιφερειών. Το SRSP συμβάλλει ενισχύοντας διοικητικές ικανότητες των κρατών μελών. Ε, η νομική βεβαιότητα και οι υψηλή ποιότητα ε, διοικητικέ υπηρεσίες ε, βελτιώνουν την, την ποιότητα της διακυβέρνησης, κάτι που με τη σειρά του ενισχύει την οικονομική ανάπτυξη στις χώρες μέλη. Οι διευθυντικές μεταρρυθμίσεις δημιουργούν ένα περιβάλλον θετικό για τις επιχειρήσεις και τους εργαζόμενους, αυξάνουν την απασχόληση και συμβάλλουν στην οικονομική και κοινωνική συνοχή. Αυτό είναι και ο λόγο που οι διαστροτικές μεταρρυθμίσει είναι σημαντικός θεμέλιος λήθος για την οικοδόμηση μια πιο ανθεκτικής ε, έγκαιρα και αποτελεσματικά τα κράτη-μέλη χρειάζεται να υπερβαίνουν εμπόδια όσον αφορά την διοικητική του ικανότητα. Και εδώ έρχεται το πρόγραμμα στήριξη διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων να συμβάλλει και είναι κάτι που το αναγνωρίζουν όλα τα κράτη-μέλη. Ήδη πριν από την έγκριση του SRSP Υπήρχε υπηρεσία ε, όπου εφηλήθηκαν από αυτό. 20 έργα στηρίξαμε, παραπάνω από τα μισά έχουν ολοκληρωθεί, κάποια ακόμη βρίσκονται υπό εξέλιξη. Επίσης ε, δόθηκε στήριξη στις σλοβενικές ε, αρχές για την αντιμετώπιση του προβλήματος των μη εξυπηρετούμενων δανείων. Όσον αφορά το πρόγραμμα στήριξης διερθών εκατομμύρια ευρώ, περίπου το 1 τέταρτο του διαθέσιμου προϋπολογισμού. 444 είναι τα ε, αιτήματα που έχουν συνολικά υποβληθεί, ε, πέντε φορές παραπάνω από τον προϋπολογισμό που έχει ε, SRSP του 2017 σε στενή συνεργασία με ε, υπηρεσίες της Κομισιόν και με τα κράτη-μέλη για να εξασφαλίσουν ότι δεν θα υπάρχει επαλήθευση. δεν θα υπάρχει επικάλυψη. Εννιά αφορούν τη στήριξη στη γραφε... στην διοίκηση άλλα ε, προ, πιστοτικό κλάδο. Συνολικά το πρόγραμμα συμβάλλει στην συνεπή ε, υλοποίηση των ε, ενωσιακών πολιτικών. 90% των πνεύματος προσαρμογής και την εφαρμογή προτεραιοτήτων όπως είναι η Ενεργειακή Ένωση, η Ένωση Κεφαλαιογορών και γενικά την υλοποίηση του Ευρωπαϊκού Δικαίου. Η παρά το γεγονό ότι το SRSP υπάρχει εδώ και 9 μήνες μόλις, ήδη έχουν βλή διαδικασία και την ε, προσαρμογή στι ανάγκε τους. Επιπλέον, οι υποστηρικτικές δραστηριότητες έχουν και μια διασυνοριακή και περιφερειακή διάσταση. Για παράδειγμα, ε, υποστηρίζουμε τις τρεις βαλτικές χώρες για την, για την ε, έναρξη εμπειριών του ενός κράτους μέλους σε άλλο κράτος μέλης. Και γενικά ε, στόχος μας είναι η ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών. Αυτό ισχύει και στα συστήματα υγείας όπου βοηθούμε στα κράτη, τα κράτη-μέλη να εφαρμόζουν τις συστάσεις αναχώρα με σκοπό να παρέχουν αποτελεσματικές και τις Ένωσης. Για παράδειγμα στη Σλοβακία δίνουμε στήριξη για την ανάπτυξη μεγαλύτερων ικανότητων για την ε, εντοπισμό επενδυτικών προγραμμάτων που μπορούν να χρηματοδοτηθούν από ευρωπαϊκά ταμεία όπως είναι το ΕΦΣΙ, σε συνδυασμό με εθνικά ταμεία και πηγές χρηματοδότησης στη Λιθουανία ε, ε, ε, ε ιδιωτικών κεφαλαίων. Ακόμη δεν έχουμε υιοθετήσει την ε, απόφαση χρηματοδότησης για φέτος, όμως μπορώ να σας δώσω κάποια πρώτα στοιχεία για την, που γενικός στόχος μας θα είναι η καλύτερη αξιοποίηση των χρηματοδοτικών μέσων και η ενίσχυση των επενδύσεων. Το χρειάζεται Ε, υπερβαίνει δυστυχώς, το ενδιαφέρον που έχει εκφραστεί υπερβαίνει δυστυχώς ε, τους ε, σημερινούς δημοσιονομικούς περιορισμούς που έχουν τεθεί. Γεγονό είναι ότι το, το σκοπός του προγράμματος είναι η ενίσχυση σύγκλησης, η υλοποίηση διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων προκειμένου λογισμού του SRSP και να ε, δημιουργηθεί ξεχωριστή γραμμή για την υποστήριξη κρατών εκτός Ευρωζώνης προκειμένου και στην πορεία τους για την ένταξη στην Ευρωζώνη. Προτείνουμε λοιπόν να ενισχυθεί το SRSP με, άλλα, ε, με επιπλέον 80 εκατομμύρια ε, ευρώ από τον Ευρωπαϊκό Προπολισμό για το κατακτήσει στην εφαρμογή των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων. Βάσει του άρθρου, βάση του άρθρου 11 του κανονισμού για το SRSP δίνεται η δυνατότητα να μεταφερθούν κονδύλια του στο SRSP. Ε, ελπίζω και το Κοινοβούλιο στην πορεία και των συζητήσεων να υποστηρίξει. Ότι το πεδίο των ερωτήσεων θα είναι ευρύ, αλλά ας ξεκινήσουμε με τους ε, εκπροσώπους των πολιτικών ομάδων. Ο κύριος Νοβάκοφ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ, κύριε Επίτροπε. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω καταρχάς που βρήκατε το χρόνο από την βεβαρημένη πιο πρόσφατη δυνατότητα που δίδεται στα κράτη-μέλη. Και αν ήταν να κάνω έναν παραλληλισμό, είναι σαν νέα για οποιοδήποτε προϊόν. Και προκειμένου να το επιτύχουμε αυτό, πρέπει να ακούμε τους πελάτες μας, που στην περίπτωση αυτή είναι τα κράτη-μέλη. Επί τη βάση λοιπόν στο βέλτιστο δυναμικό. Έχοντας λοιπόν εντοπίσει αυτό το μειονέκτημα δηλαδή και έχουν καταβληθεί πολύ σημαντικές προσπάθειες και υπάρχει ενδιαφέρον που έχει εκδηλωθεί. Είχαμε ξεκινήσει με μια υπόσχεση προς τα κράτη-μέλη για ένα αποθεματικό επίδοσης. Και τώρα κάπου καιρό εδώ στο Κοινοβούλιο και στην Επιτροπή Προεπολογισμού ακούω τους συναδέλφους της Επιτροπής εκείνης τη δυνατότητα της ευελιξίας χρησιμοποίησης αυτού του μέσου, ότι δηλαδή λένε ότι αυτή η ευελιξία είναι πολύ περιορισμένη. Και εκπλήσωμε του μέσου ευελιξίας, ωραία το έχουμε αυτό η διάθεσή μας. Εάν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί να μας πει ότι έχουμε περιθώρια και εξεπλάγει που άκουσα ότι ακόμα και 24 κράτη-μέλη συμμετέχουν. Όρους για τα ερχόμενα δύο έτη, αλλά αυτό μέσω του μέσω ευελιξίας. Δεν μπορούμε να αφαιρέσουμε, να μεταφέρουμε από την πολιτισμό. Είναι σε θέση να προτείνουν και έργα μεταρρύθμισης Και μάλλον το καθήκον των ε, μελών του Κοινοβουλίου δεν είναι να κάνουμε καλή ε, δουλειά για το Γιούγκερ. Έχουμε το Ταμείο Συνοχής για την Ευρωζώνη, έχουμε τις ε, δυνατότητες μεταρρυθμίσεων ήδη εντός. Είναι οι περιφερειακές. Και το έχουμε συζητήσει όταν ξεκινήσαμε με το SRSP για το πώς θα λύσουμε ό,τι αντιθέσεις υπάρχουν με το, μεταξύ του εθνικού επίπεδου και του περιφερειακού επίπεδου. Πώς θα χρησιμοποιήσουμε ότι αντιθέσεις υπάρχουν με το, μεταξύ του εθνικού επίπεδου και του περιφερειακού επίπεδου. Πώς θα χρησιμοποιηθεί αυτή η χρηματοδότηση. Εσείς βλέπετε ότι όντως υπάρχει κάποια σύγκρουση εδώ. Και πώς θα διασφαλίσουμε ότι δεν θα γίνουν προτάσεις ανεξάρτητα Πώς βλέπετε εσείς να λειτουργεί το SRSP με τις προτάσεις για επιδόσεις και πώς νομίζετε ότι θα γίνει η εφαρμογή τα επόμενα χρόνια. Ευχαριστώ πολύ. Αν δεν υπάρχουν άλλες ερωτήσεις, το λόγο έχει ο Επίτροπος για να απαντήσει. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ για τις ερωτήσεις αυτές και τα σχόλιά σας. Ποιή κατά 80 εκατομμύρια ευρώ. Από εκεί και πέρα υπάρχουν και διάφορες άλλες ξεχωριστές προτάσεις που αφορούν σχετικά με τις μεταρρυθμίσει μετά το 2020 και τις προτεραιότητες στην ανακοίνωση για το ΠΔΠ που παρουσιάσαμε την προηγούμενη εβδομάδα. Το SRSS και το SRSP είναι θέματα για τα οποία εγώ είμαι ο κύριος υπεύθυνο για το, για το MFF ξέρετε ότι είναι υπεύθυνο που έχουν τεθεί σήμερα τα ερωτήματα που αφορούν την, το πρόγραμμα στήριξη διαχρονικών μεταρρυθμίσεων και την πρότασή μα να αυξηθεί ο προπολογισμό αυτού του προγράμματο. Το σκεπτικό λοιπόν είναι σαφέ και είναι το εξή. Η ζήτηση από τα κράτη-μέλη υπερβαίνει κατά πολλέ φορέ τα διαθέσιμα κονδύλια, ότι υπάρχει ανάγκη να αυξηθεί η στήριξη. Βεβαίως το ερώτημα είναι από πού θα προέλθουν τα χρήματα. Και είναι εύλογο το ερώτημα αυτό. Εδώ προτείνουμε να χρησιμοποιήσουμε το μέσο 2020. Για το ερώτημα που αφορούσε το συνολικό ύψος του προπολογισμού,